Και σημαίνει επίση ότι πρέπει να αποφασίσουμε πού θα γίνουν οι επενδύσει για να έχουμε τη μεγαλύτερη επίπτωση στην καθημερινότητα των Ιταλών και των άλλων Ευρωπαίων. Γι' αυτό, τον περασμένο Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε έναν δίκαιο και ισορροπημένο προπολογισμό για το μέλλον, που είναι πιο αποτελεσματικό και εστιάζει περισσότερο στα θέματα που ενδιαφέρουν και θίγουν του περισσότερου συμπολίτε μα. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τριπλασιασμό των πόρων για την μετανάστευση και την ασφάλεια. Σχεδόν τριπλασιασμό. Σχεδόν 33 δις. Και πρότεινε έναν πιο αποτελεσματικό προϋπολογισμό για την εξωτερική δράση, για να φτιάξουμε συνεργασία με τις χώρες στη γειτονία μας και ευρύτερα. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ιταλία, που είναι χώρα που έχει αναλάβει τόση ευθύνη για τα θέματα αυτά θα επενδύσουμε ούτω ώστε η οικονομία μας να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο καινοτόμα, πιο παραγωγική. Και κλειδί για την Ιταλία θα είναι το 50% αύξηση στην χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία και τα 9 δις για την ε, ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία για να γίνει στην Ιταλία η ψηφιακή μετάβαση. Η επένδυση στο μέλλον σημαίνει επίση να επενδύσουμε και στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή πρότεινε διπλασιασμό του προπολογισμού σε 30 δις για το πρόγραμμα Erasmus ΣΥΝ που είναι σύμβολο για την κινητικότητα της Ένωσης. Θέλουμε να αυξήσουμε τη στήριξη σε όλους τους τομείς και για την ανώτερη εκπαίδευση και για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το 2017 πάνω από 65.000 Ιταλοί συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα οικοδομήσει περαιτέρω επί των επιτυχιών του ε, προγράμματος Juncker. Η Ιταλία είναι μία από τους ε, δικαιούχους που έλαβε τα περισσότερα ποσά, πάνω κάτω 58 δις, που βοήθησαν την Ιταλική οικονομία και πάνω από 2.015 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν χρηματοδοτήσεις. Το σχέδιο Juncker έχει αυξήσει κατά πολύ τι ιδιωτικέ αλλά και τι δημόσιε επενδύσει στην Ιταλία. Είναι θετικό σήμα γιατί δεν πρέπει να ε, πληρώνει πολύ ο φορολογούμενο αν μπορούμε να κινητοποιήσουμε ιδιωτικέ επενδύσει. Έτσι σημειώνεται διαφορά παντού στην Ιταλία. 70 εκατομμύρια ευρώ βοηθάνε να ανακαινιστεί το νοσοκομείο του Τρεπίζο. 200 εκατομμύρια θα βοηθήσουν το Ιντερνετικό δίκτυο και θα δώσουν κατάρτιση ε, στη χρήση του Ιντερνετ σε 4 εκατομμύρια. Και 500 εκατομμύρια θα βοηθήσουν γενικότερα, ούτως ώστε 7 εκατομμύρια στην Ιταλία να έχουν ευρυζωνική σύνδεση. 7 εκατομμύρια νοικοκυριά. Και το πρόγραμμα InvestEU μπορεί να κάνει ακόμη πολύ περισσότερα. Συνολικά θέλει να μοχλεύσει 650 δις επενδύσεων. Όλα αυτά μπορούν και θα σημειώσουν ουσιώδη διαφορά και πρόοδο στην Ιταλία, επιτόπου και παντού στην Ένωση. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν είναι δύσκολο να υπάρξει ανάπτυξη σε πολλές χώρες, γιατί υπάρχουν ε, παγκόσμιες αβεβαιότητες αλλά και σε ορισμένες και λόγω εγχωρίων ε, αποφάσεων. Για να υπάρξει ανάπτυξη χρειάζεται εμπιστοσύνη και στα νοικοκυριά και στους επενδυτές η ε, εμπιστοσύνη είναι στο, σαν το οξυγόνο. Αντιλαμβάνεσαι ε, ότι υπάρχει μόνο όταν ε, δεν υπάρχει επαρκέ και αν δεν υπάρχει επαρκή εμπιστοσύνη δεν γίνονται οι αναγκαίες επενδύσεις. Η επένδυση στην Ιταλία είναι πιο αδύναμη από το μέσο όρο τη Ένωση για πολλά χρόνια. Και αυτό είναι διαθωτικό πρόβλημα και δημιουργεί λιγότερε θέσει απασχόληση για του Ιταλού. Παράλληλα, όπω επανειλημμένα λέω, η Ιταλία είναι μεταξύ των πιο δημιουργικών οικονομιών στον κόσμο. Το μέλλον της χώρας σας είναι στα χέρια σας. Να κάνετε αυτό που είναι αναγκαίο για να αποδεσμευτεί αυτή η δημιουργικότητα και να δώσετε ένα περήφανο μέλλον στους Ιταλούς. Κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμοι βουλευτές, περάσαν δύο χρόνια από τότε που υποβάλαμε το... τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης, που ξεκίνησε τη συζήτηση που διεξάγεται τώρα για το τι θέλουμε να επιτύχει η Ένωσή μας τα επόμενα χρόνια. Πέντε εναλλακτικέ λύσει έδιναν ε, πέντε διαφορετικέ πορείε από τον οποίο μπορούσαμε να ε, αποφασίσουμε. Αλλά ό,τι και να επιλέξουμε, ορισμένα θέματα είναι σταθερέ. Και ένα από αυτά είναι ο κεντρικό ρόλο τη Ιταλία στην περαιτέρω πορεία τη Ένωση. Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Ιταλία. Και η Ιταλία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη. Δεν είναι έκπληξη, ούτε σύμπτωση που οι πρώτε γραμμές της Λευκής Βίβλου ήταν για τον Σπινέλη και τον Ρώση και το μανιφέστο τους. Οπότε, οδεύοντας προς το μέλλον, πρέπει να εμπνεώμεθα όλοι από τους προκατόχους μας για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή, πιο ενωμένη ένωση για τις επόμενες γενναίες. Όπως έκανε και εκείνη για μας, ευχαριστώ πολύ. Τώρα προχωρούμε στις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Βέμπερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξεκινήσατε από την προοπτική του λαού. Εγώ είμαι τη Βαβαρία. Πηγαίνω στις εκκλησίες, στην εκκλησία, στα, στο νοσοκομείο, στο δρόμο, μιλώ με τους ανθρώπους και διαπιστώνω τα ίδια προβλήματα που αναφέρετε. Κοινωνική δικαιοσύνη, οι προοπτικές για τους νέους. Για να απαντήσουμε πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι πέραν αυτών που μας είπατε. Για να απαντήσουμε στα οικονομικά προβλήματα η Ιταλία, πρέπει να πούμε ότι η Ιταλία έχει σήμερα, είναι η χώρα με το μικρότερο ρυθμό ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα για την Ιταλία. Είναι πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για την... Ε, είστε χώρα της ομάδας των 7, μια, μια κινητήρια δύναμη στην Ευρώπη. Τι πρέπει να κάνουμε. Στο ΕΛΚ πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις. Και είδαμε ότι η κυβέρνηση στην Ιταλία δεν συμφωνεί ούτε καν για την ολοκλήρωση ενός ήδη εγκεκριμένου έργου μεταξύ Γαλλίας, ε, Γαλλίας Ιταλίας η κυβέρνησή σας για εβδομάδες ε, στο ξεκίνημά σας συζητούσε για το αν θέλετε ή όχι να είστε μέλη στην Ευρωζώνη. Πιστεύουμε ότι μόνο με μεταρρυθμίσεις μπορούμε να χτίσουμε το οικονομικό μέλος, μέλλον της χώρας σας. Και αυτό δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά και άλλες ε, χώρες που ή στην Κύπρο, στην Ισπανία, στην Ελλάδα είδαμε ότι αν θέλεις μπορείς να αλλάξεις την αγορά εργασία, το δικαστικό σύστημα, το φορολογικό σύστημα για να δώσεις θέσεις εργασία. Και στη Γερμανία τη χώρα μου η Ατζέντα 2010 του, του κυρίου Σρέντερ θεμελίωσε την μεταρρύθμιση. Μεταρρυθμίσεις λοιπόν για το μέλλον. Στην κυβέρνησή σας η κυβέρνηση δεν, δεν προσβλέπει στο μέλλον. Επίσης θεωρούμε ότι ένας σταθερός προπολογισμό είναι κρίσιμος για μια ισχυρή οικονομία, κάτι που δεν βλέπουμε στην Ιταλία. Αυξάνεται το χρέος, αυτό βλέπουμε. Αυτά συνοπτικά. Οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιταλία επιπλέον είναι πρόβλημα. Υπάρχει έλλειψη ανάπτυξης στην Ιταλία και είναι ευθύνη όχι της Ευρώπης αλλά της Ιταλικής κυβέρνησης. Εμείς σεβόμαστε απόλυτα το ότι είσαστε μια δημοκρατική κυβέρνηση με εντολή από τους ψηφοφόρους σας. Είναι ευκολότερο ίσως να κερδίσει εκλογές ως ένα κίνημα κατά τον ελίτ από το να μείνει στην κυβέρνηση ως ένα κίνημα κατά τον ελίτ. Κάποιοι γίνατε ή φτάσατε να γίνετε νέες ελίτ μετά στην Ιταλία. Να υπογραμμίσω ένα δεύτερο θέμα για το, μεταν, για το μεταναστευτικό, το ΕΛΚ πιστεύει ότι η Ιταλία αξίζει την αλληλεγγύη της Ευρώπης, κατανοεί την οργή των πολιτών της Ιταλίας. Για πολλά χρόνια η Ιταλία ήταν μόνη της και γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε ένα μηχανισμό αλληλεγγύη για την, αλληλεγγύης για την Ένωση, αλλά είναι πρόβλημα για μας να βλέπουμε ότι ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έρχεται εδώ και μας λέει ότι το όργανο στο οποίο μετέχει δεν ε, υλοποιεί τις υποσχέσεις του. Εσείς πρέπει να το κάνετε αυτό. Για τις εξωτερικές σχέσεις, να σας ευχαριστήσω που υπογραμμίσατε την ευρωπαϊκή μας προσέγγιση ε, στην απάντησή μας για τη Ρωσία. Η Ιταλική κυβέρνηση περιμένουμε να συνενέσει στις κυρώσεις. Από την άλλη, τις τελευταίες μέρες είδαμε τις συζητήσεις για την Βενεζουέλα. Για το ΕΛΚ έχουμε εκεί έναν δικτάτορα ο οποίος έφτασε στην έγινε στην εξουσία με αντιδημοκρατικές εκλογές, με τη βοήθεια του στρατού που εμποδίζει ακόμα και τη μεταφορά φαρμάκων στη χώρα του. Και απ' την άλλη έχουμε ένα ελεύθερο εκλεγμένο κοινοβούλιο που ζητά απλά το δικαίωμα να γίνουν νέες πρόορες εκλογές για τη θέση του Πρόεδρου. Σε μια επιστολή που έστειλε σήμερα προς τους Ιταλούς πολίτες, ο κ. Γκουαϊντό ρώτησε γιατί η Ιταλική κυβέρνηση δεν, υποστηρίζει, δεν υποστηρίζει τις δημοκρατικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα. Θα πρέπει να απαντήσετε σε, αυτό, σε αυτή την επιστολή αν πιστεύετε σε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής κάποιες γενικότερες ε, σκέψεις. Ευχαριστώ για την δέσμευσή σας να αναζητήσετε κοινέ ευρωπαϊκές λύσεις. Είπατε σήμερα ότι η Ιταλία γίνεται πιο παρούσα, πιο φωνάζει περισσότερο στην στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η δυνατή φωνή στην ευρωπαϊκή συζήτηση μπορεί να δείχνει εγωισμό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι βούληση συνένεσης, γιατί αν φωνάζουν όλοι, μόνο θόρυβος γίνεται. Είπατε επίσης για την ανάγκη να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ λαού και ευρωπαϊκών θεσμών. Είστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι όλοι εδώ, η Λέγκα, ε, τα Πέντε Αστέρια, το, το Δημοκρατικό Κόμμα, Όλοι είμαστε εδώ, όλοι είμαστε ε, εκπρόσωποι των πολιτών, δεν είμαστε η ελίτ. Εδώ είμαστε εκπρόσωποι των λαών και εδώ πρέπει να αποφασίσουμε για το μέλλον. Ευχαριστώ. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες το λόγο έχει ο πρόεδρος Ούντο Μπούλμαν. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα που ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ είναι το σπίτι της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Ένας χώρος δημόσιας συζήτησης και ειλικρίνειας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ειλικρινείς δηλώσεις και να σας ε, ενημερώσω για τις ανησυχίες μου. Ανησυχώ όταν ε, η κυβέρνηση μιας συντηρητικής χώρας και η κυβέρνηση της 7ης βιομηχανικής δύναμης στον κόσμο οδηγεί το Ιταλικό έθνος όλο και πιο πολύ σε οικονομική και πολιτική απομόνωση. Αυτό γίνεται σήμερα. Ενώ έχουμε ένα πλαίσιο, μια εξωτερική συγκυρία, όπου από τη μία δεν μπορούμε πλέον να βασιστούμε στην Ουάσιγκτον όπως το παρελθόν και αντιμετωπίζουμε και νέες απειλές από τη Ρωσία. Η οικονομία σας οδεύει προς την ύφεση και βλέπουμε ότι η βιομηχανική σας παραγωγή πέφτει. Σε αυτή την κατάσταση λυπάμαι ιδιαίτερα από την ε, ε, άνευ νοήματος κλιμάκωση των εντάσσεων μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας. Μα τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, σε τι χρησιμεύουν. Γιατί δημιουργείτε συγκρούσεις κάτι τέτοιο, το ξέρετε, κανείς δεν κερδίζει από τέτοιες συγκρούσεις. είναι μια κατάσταση όπου όλοι θα χάσουν. Και η χώρα σα και η Ευρώπη. Ο πληθυσμό και των δύο χωρών μπορεί να πληρώσει υψηλή τιμή. Η Ιταλία και η Γαλλία είναι ο καθένα ο δεύτερο εμπορικό εταίρο του άλλου. 17,6 δι είναι το ύψο του, ε, ε, ε, του ετησίου εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Εκατοντάδε χιλιάδε θέσει εργασία εξαρτώνται. Και αυτέ οι θέσει εργασία δεν είναι των ελίτ. Είναι απλών ανθρώπων και ο Ιταλικός λαός ε, δεν μπορεί να χάσει περισσότερο θέσεις εργασίας. Η Ιταλία φέτος θα αυξηθεί μόνο κατά 0,8%. 0,8%. Το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Μπορείτε να τα παρουσιάζετε αυτά ε, λέγοντας ότι θέλετε να επανέλθει η αξιοπρέπεια της εργασίας. Ε, δεν βλέπω όμως να οδεύεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν βλέπω να επανέρχεται η αξιοπρέπεια της εργασίας. 75.000 ε, εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους και πολύ περισσότεροι είναι σε επισφαλής και χαμηλόμιστες εργασίες ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εγκαταλείπουν τη χώρα σας ψάχνοντας για μια καλύτερη ζωή και σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά οι οικονομίες των Ιταλικών οικογενειών τέθησαν εν κινδύνων με μία, λόγω μιας εσκεμμένης αντιπαράθεσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προπολογισμό σα. Ήταν αναγκαίο αυτό. Ή ήταν μόνο μία προσπάθεια προπαγάνδας ενός και μόνο ανθρώπου. Αυτό κόστισε στους Ιταλούς 1,7 δις μόνο κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών. Και γιατί, ούτω ώστε ο Σαλβίνη να έρχεται και να κάνει φιγούρα στι Βρυξέλλε. Ο οποίο έχει έναν αποδιοπημένο τράγο για όλου. Αλλά καμία λύση για τίποτα. Αυτή είναι σήμερα η Ιταλική πραγματικότητα. Από αυτό το οικονομικό χάος ο Σαλβίνη τώρα προσπαθεί να αξιοποιήσει την ε, μετανάστευση. Ήμουν πριν από δύο εβδομάδες στην Κατάνια και εκεί είδα ότι 47 άτομα, 47 άτομα για 12 μέρες δεν μπορούσαν να βγουν από το σκάφος που τους είχε διασώσει το Sea-Watch. Μεταξύ αυτών ήταν και ανήλικοι και θύματα βασανιστήριων. Γιατί, γιατί, γιατί είχαν γίνει παιχνιδάκι μια κοινική πολιτικής. Αυτή δεν είναι η Ιταλία που ξέρουμε, συνάδελφοι. Γνωρίζουμε μια άλλη Ιταλία. Ξέρουμε τη μεγάλη ευρωπαϊκή Ιταλία του Αλτιέρο Σπινέλη του Ντεγκάσπερη που ποτέ ποτέ για μικροπολιτικό υποτιθέμενο κέρδος δεν ε, ε, έθεσαν εν κινδύνο την Ευρώπη ούτε τη χώρα τους. Καταλαβαίνω πολύ καλά και η ομάδα μου καταλαβαίνει πολύ καλά γιατί είναι απογοητευμένοι πολλοί πολίτες στην Ιταλία. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχε επιτύχει πολλά πράγματα είχε σώσει χιλιάδες και χιλιάδες από πνιγμό στη θάλασσα και η Ευρώπη δεν σας βοήθησε αρκετά. Δεν σας ε, επέδειξε επαρκή αλληλεγγύη. Αλλά ποιος σας απογοήτευσε. Όχι οι φιλοευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Όχι εκείνοι που θέλουν να προωθηθεί η Ευρώπη. Κοιτάξτε. Πείτε στους πολίτες σας ποιος δεν σας βοηθάει να κάνετε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Είναι οι φίλοι του κυρίου Σαλβίνη. Είναι οι Κατσίνσκι και οι Όρμπαν και ο, ο Κούρτ στην Αυστρία. Αυτοί τα μπλοκάρουν όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πείτε την αλήθεια. Ενώ οι φιλοευρωπαίοι πάντα είναι στο πλευρό σας. Όταν ε, σώζετε ανθρώπους στη θάλασσα. Και είναι λογικό βέβαια αυτό να το κάνει. Υπάρχει ακόμη αυτή η Ευρώπη. Υπάρχει ακόμη αυτή η Ιταλία. Και οι δύο αγωνίζονται αυτή η θαυμάσια Ιταλία, αυτό το θαυμάσιο έθνος. Η Ιταλία του Σπινέλη και του Ντεγκάσπερη. Αυτό βλέπω όταν βλέπω τους ψαράδες της Λαμπεντούζα που παρά τους νόμους Μπόση Φίνη ενώ ξέρανε τους περίμενε παρόλα αυτά συνέχισαν να σώζουν ανθρώπους στη θάλασσα. Το βλέπω στους ε, ε ναυτικούς του Ντετζότη που είναι ένα ε, σκάφος της Ιταλικής ακτοφυλακής που δεν έπρεπε να το κάνουν αλλά παρόλα αυτά είπαν ότι έχουμε έναν κώδικα δεντολογίας ε, των ναυτικών και το κάναμε και το βλέπουμε αυτά στους ε, δημάρχους που δίνουν κατάλημα και τροφή στους πρόσφυγες ακόμη και αν το αρνείται η κυβέρνηση αυτοί διασώζουν την αξιοπρέπεια της Ιταλίας αυτή είναι η τεράστια η θαυμάσια Ιταλία των ευρωπαϊκών αξιών αυτή την Ιταλία θαυμάζουμε σε αυτήν απλώνουμε το χέρι γιατί χρειαζόμαστε αλλά τότε θα πρέπει να σταματήσει η κυβέρνησή τους να φοράει αυτή τη μάσκα της απαθροπιάς. Γιατί αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική Ιταλία. Πρέπει επιπλέον να ξυπνήσει η, Ιταλία κατά τον η Ευρώπη κατά των λαϊκισμών, κατά αυτών που καταστρέφουν τις πατρίδες μας. Στην Ιταλία αξίζει η αλληλεγγύη μας. Η Ιταλία είναι στην καρδιά της Ευρώπης. Μαζί με τους στενότερους φίλους της. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Φίτο που θα μιλήσει από το ECR, θα ήθελα να πω στου ε, ε, εκπροσώπους πολιτικών ομάδων ότι αν υπερβαίνουν το χρόνο τους τον ε, μειώνουν από τους ομιλητές, από τους ανεξάρτητους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Και όπως ξέρετε πρόκειται για μια χώρα που έχει κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Σε αυτό έχουν αναφερθεί πολύ. Ε, δεν έχει νόημα να κάνουμε μία γενική συζήτηση. Πολλές φορές οι διαγνώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με την απτή πραγματικότητα. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να σταθώ στις επικρίσεις για το τι αποτελεί, τι από τι απαρτίζεται η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια σε, στον οικονομικό τομέα, στο μεταναστευτικό και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό να δώσουμε ορισμένα στοιχεία σαφήνειας με συγκεκριμένα παραδείγματα, αντιφάσεις, τις οποίες θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Γιατί όταν μιλάμε για μετανάστευση, και τη στιγμή που η κυβέρνησή σας κατά αυτή τη θητεία προέβαλε μία δράση όχι τόσο αρνητική, αλλά που προσπάθησε να βρει λύσεις σε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους ε, ψαράδες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι όχι μόνο σώζουν ζωές, αλλά διαμαρτύρονται για θέματα που τους αφορούν εξαιτίας των πολιτικών μας. Ως προς το μεταναστευτικό, συμφωνούμε, αλλά τι θα γίνει με το σύμφωνο σταθερότητας. Εδώ υπάρχει μεγάλη ε, ανασφάλεια. Μιλήσατε στα Ηνωμένα Έθνη, ε, μιλήσατε για τη διάσκεψη του Μαρακές μετά στηρίσατε στάση αποχής για τη Βενεζουέλα. Μιλήσατε για ενιαία φωνή, αλλά στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών ε, εξαιτίας της αρνητικής ψήφου της Ιταλίας δεν μίλησε η Ευρώπη με μία φωνή στα οικονομικά. Έχετε δίκιο ως προς την ανάλυση σας, αλλά τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματά σας είναι λανθασμένα. Δεν υπάρχουν επιλογές διαρθρωτικών πολιτικών. Αντίθετα, πολλοί λένε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος αύξησης του ελλείμματος. Εμείς το αυξάνουμε γιατί υπάρχουν πολιτικές που επιβαρύνουν τις δημόσιες δαπάνες. Μην μιλάμε ε, λοιπόν για διαρθρωτικές ε, αλλαγές. Σήμερα ζούμε δύσκολες στιγμές. Σήμερα μας μιλάτε για την ανάπτυξη και το ρόλο της Ιταλίας. Ο Υπουργός ε, Υποδομών σας θέλει να μας δείξει ότι το ΤΑΒ είναι ένα μεγάλο λάθος και θα πρέπει να μπλοκαριστεί. Πρόκειται για την γνωστή σιδηροδρομική γραμμή. Γι' αυτό θα πρέπει τα συμπεράσματά σας να οδηγήσουν στην πράξη. Και δυστυχώς η πράξη δεν οδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση ούτε για την Ιταλία ούτε για την Ευρώπη. Από πλευράς ελευθέρων το λόγο έχει ο Γκί Φερχόφστατ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω Ιταλικά, Πρόεδρε. Γιατί πέραν της χώρας μου, μάλλον, κύριε Κόντε, είμαι ερωτευμένος με την Ιταλία και με τους Ιταλούς. Για μένα, η Ιταλία δεν είναι χώρα, είναι πολιτισμός. Είναι εκεί όπου γεννήθηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και για αιώνες συγγραφείς, καλλιτέχνες, διανοούμενοι επισκέπτονταν την Ιταλία τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους για να ανακαλύψουν την Ιταλία το να ανακαλύψουν την Ιταλία σημαίνει να επισκεφθούν την Ιταλία να πάνε στη Φλωριντία, στη Ρώμη, στη Νάπολη. Ε, Μοντένια Λαφάτο. Για να πεθάνουν. Ο Γκέτε αυτό έκανε. Και γι' αυτό, κύριε Κόντε, με πονάει, κύριε Κόντε, που βλέπω σήμερα την ε, πολιτική αποδυνάμωση της Ιταλίας. Κάτι που δεν ξεκίνησε πέρσι, πριν από ένα χρόνια, πριν από 20 θα έλεγα. Η εντύπωσή μου είναι ότι η πανέμορφη αυτή χώρασε, πέρασε από το να είναι ένας από τους ιδρυτές της Ευρώπης και ένας από τους ε, υποστηρικτές της Ευρώπης στον τελευταίο τροχό. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω και εγώ και το Κοινοβούλιο και ο εξωκόσμος. Και αυτό δεν ξεκίνησε με τον Πρωθυπουργό Κόντε. Ξεκίνησε με την ε, κακή διακυβέρνηση της εποχής Μπερλουσκόνη και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το Μαλ αυτή η κακή διακυβέρνηση, επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας από τον Σαλβίνη, από τον Τιμάιο, τους πραγματικούς ηγέτες αυτής της κυβέρνησης μιας κυβέρνησης με συμπεριφορά μερικές φορές κύριε Κόντε αντιευρωπαϊκή και μερικές φορές με συμπεριφορά που έδειχνε μίσος κατά άλλων κρατών μελών, μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας. Και η Ιταλική κυβέρνηση, η Ιταλική κυβέρνηση είναι αυτή που ε, εμπόδισε την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί ενωμένη απέναντι στο Μαδούρο και να αναγνωρίσει τον Γκουαϊντό ε, προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας. Και το ξέρετε. Γιατί. Γιατί το κάνατε. Το κάνατε κάτω από την πίεση, πίεση του Κρεμλίνου, του Πούτιν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό μίλησε κάποιος γι' αυτό ήδη. Πρέπει να σταματήσουμε τον κανόνα ομοφωνία στο Συμβούλιο, το συντομότερο δυνατό η Ιταλική κυβέρνηση δεν μετέχει στην πλειοψηφία του Συμβουλίου στην αλλαγή της ε, πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης. Ο κ. Σαλβίνη θέλει να μπλοκάρει τα λιμάνια, ε, την είσοδο στα λιμάνια των μεταναστών, αλλά ταυτόχρονα μπλοκάρει την ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα, την μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Και για μένα αυτό είναι παράλογο, μια παράλογη συμπεριφορά, γιατί οι Ιταλοί πολίτες είναι οι πρώτοι που πληρώνουν την έλλειψη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα αυτό. Αυτό είναι το τρίτο παράδειγμα που θα δώσω. Τον τελευταίο χρόνο εσείς, η κυβέρνησή σας, είστε υπεύθυνοι για την στασιμότητα και φοβάμαι αύριο την ύφεση της Ιταλικής και Ευρωπαϊκής οικονομίας. Η κυβέρνησή σας έχει μόνο μία τακτική να ε, επανεκλεγεί κάνοντας δώρο χρέος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η τελευταία ελαφρότητα της κυβέρνησής σας, της κυβέρνησης από πλευράς Ντιμάιο που εκμεταλλεύεται τη θέση του για να υποστηρίξει τα ζηλέ ζών, τα κίτρινα γυλαίκα, ένα λαϊκιστικό ε, μοντέλο που υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι που καίνε αυτοκίνητα, κλέβουν ε, μαγαζιά και καταστρέφουν στάσεις λεωφορείων. Ο Ντιμάιο συνάντησε τον Κριστόφ Σαλανσό. ο οποίος ζήτησε δύο φορές να γίνει πραξικόπημα κατά του εκλεγμένου Προέδρου της Γαλλικής ε, Δημοκρατίας. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Αυτό είναι μία ανεύθυνη συμπεριφορά. Όχι συμπεριφορά ενός αντιπροέδρου της κυβέρνησης μιας μεγάλης κοινοτικής χώρας. Πριν από ένα χρόνο, ίσως θυμάστε, στις 23 Νοεμβρίου του 2017, ο κύριος Δημάιο είχε στείλει μια ανοιχτή επιστολή στον Εμμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας το θαυμασμό του και πρότεινε το κίνημα, ότι το κίνημα των πέντε αστέρων ήταν ε, η, ιταλική εκδοχή του Αν Μάρς. Γελία συμπεριφορά. Η ερώτησή μου προς εσάς κύριε Πρωθυπουργέ είναι για πόσο καιρό θα είστε ο, ο χειράνθρωπος του Ντιμάιο και του Σαλβίνη. Σας καλώ σε κάτι εμπνευστείτε από τους λαμπρούς Ιταλικούς, Ιταλούς συμπατριώτες σας. Σπινέλη, Τσιάμπη, Ναπολιτάνο, Ντράγκη, ναι, ναι. Το Τζότζιο Ναπολιτάνο, ναι. Ένα μεγάλο Ευρωπαίο με πραγματική ιδέα και μεγάλο άνθρωπο σε, αυτό το σώμα. Και μην ξεχάσετε τη φίλη μου Εμπαμπονίνο. Αυτοί είναι οι άνδρες και οι γυναίκες που είναι το μεγαλείο της Ιταλίας και που έπαιξαν ένα μεγάλο ρόλο στην Ευρώπη. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του κυρίου Κόντε και όλων αυτών των προσωπικότητων που ανέφερα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους ευρωβουλευτές ότι εδώ δεν είμαστε στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Ε, μιλάμε για τις ευρωπαϊκές προοπτικές και συζητάμε τις προτάσεις της Ιταλίας ως προς την ευρωπαϊκή προοπτική. Το πολιτικό μου δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση Κόντε. Απλώς θέλω να έχουμε μία συζήτηση που να μην αφορά την κατάσταση στην Ιταλία. Γιατί δεν είναι αυτό το θέμα της συζήτησης. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά σας λέω ποιος είναι ο στόχος της συζήτησης. Λοιπόν, η κυρία Φορέντσα από την ΚΟΕ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ΚΟΕ θα ήθελα να υποβάλω ορισμένα ερωτήματα προς τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας ως προς το τι θα συμβεί, τι συμβαίνει και τι θα συμβεί στην Ιταλία. Δυστυχώς οι συνέπειες θα είναι πάντα ολέθριες, νεοφιλελεύθερες ε, πολιτικές και ένα μεγάλο κύμα αντίδρασης και με τις δύο επιλογές φτάνουμε σε ολέθρια αποτελέσματα. Ε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τους πληθυσμούς, τις γυναίκες, τους άνδρες, τη δυνατότητα δράσης, να καταπολεμήσουμε και να ε, ρίξουμε τα δεσμά του νεοφιλελευθερισμού. Να μιλάμε για ισότητα, γιατί μας πρόδωσε αυτή η κυβέρνηση. Δυστυχώς ε, η σχέση ελίματος ΑΕΠ επιδεινώθηκε και ως προς το ίσο εμπόριο, ίσον όρον εμπόριο, δεν υπάρχει θέση της Ιταλικής κυβέρνησης για τη ΣΥΤΑ. Και νομίζω ότι η Ιταλική κυβέρνηση θέλει να φτάσει σε ε, ένα, ε, μια διαφορετική αντιμετώπιση των πλουσίων. Θα πρέπει να δώσετε μία απάντηση και γιατί με μεσημβρινή ε, Ιταλία. Επίσης, ως προς τον φυσικό αγωγό, τον διατλαντικό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μία ισότητα, να μην προσφέρουμε δωρεάν εργασία που πλήττουν την αξιοπρέπεια των Ιταλών. Η Oxfam μας δίνει απτά στοιχεία. Εσείς επιβάλλετε ένα flat tax, δηλαδή έναν καταποκοπή φόρο ανεξάρτητα από το εισόδημα. Μα αυτό είναι ο νέο φιλελευθερισμός και δεν μας απασχολεί μόνο αυτή η πτυχή του ζητήματος. Στις 25 Οκτωβρίου 2018, μετά από ε, μία επίθεση της Casa Pound στο Μπάρι, απαγορεύτηκε οι νεοναζιστές και νεοφασίστες να μπορούν να δρουν έτσι δημοσία πώς θα συνδράμετε στην εφαρμογή αυτού του διατάγματος και πώς βλέπετε τις σχέσεις του Υπουργού Εσωτερικών και των ε, εκπροσώπων της Casa Pound, που είναι ένα σχήμα νεοφασιστών και τίποτα άλλο. Η Χάνα Άρεντ μας το δίδαξε αυτό. Αυτή είναι η ρίζα της κακοδαιμονίας. Αυτός είναι ο φασισμός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο Open Arms όταν διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπαμε ότι δεν μπορείτε να δράτε έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Τα λιμάνια έκλεισαν για τα για τους 59 ανθρώπους που βρίσκονταν στην ανοιχτή θάλασσα. Τι κάνατε, τι κάνετε με την Τουρκία, δεν κάνατε τίποτα. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου και υποχρεωτική relocation. Εσείς τι κάνετε. Επίσης, η ΜΚΟ δρούν στη θάλασσα. Εσείς στην ουσία τι κάνετε, κρίνετε τις ΜΚΟ και τους αντιμετωπίζετε ως εγκληματίες, δηλαδή στην ουσία εξισούνται οι ΜΚΟ με τους διακινητές. Αυτό κάνετε. Η Άντα Κολάου, όπως και η Άντα Κολάου, θα ήθελα να σταματήσετε αυτή την ολέθρια πολιτική κλεισίματος των ε, λιμανιών και η δίωξη των ΜΚΟ. Τι μπορείτε να πείτε εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον της, αν ακολουθείτε μία τέτοια πολιτική κατά των ε, μεταναστών. Στις 8 Μαρτίου θα δράσουν οι γυναίκες, οι φεμινίστριες, θα κατεβούν στις πλατείες, γιατί όταν αυτή η κυβέρνηση μιλά για τα δικαιώματα των ε, γυναικών, κάνει το αντίθετο. Μία αντιπροσωπεία της Επιτροπής ΦΑΜ βρέθηκε στην Ιταλία γιατί είδαμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να λάβουν το, χώρο, το λόγο οι γυναίκες. Τι γίνεται για τις ε, ε, γυναίκες, με τις γυναίκες της Ρώμης. Τι γίνεται με το Λουίτζι Σιέστα, τι γίνεται με το σχέδιο κατά της βίας, τι γίνεται με τον ελάχιστο ευρωπαϊκό μισθό. Έτσι θα μπορέσει να επαναξεκινήσει το μέλλον της Ευρώπης. Για να σώσουμε την Ευρώπη από το ναυάγιό της, θα πρέπει να έρθουμε αντίθετοι σε αυτές τις πολιτικές, αλλά και την πολιτική της κυβέρνησής σας. Σας παρακαλώ να μιλάτε πιο αργά, αν θέλετε να σας παρακολουθούμε, γιατί δυσχεραίνεται το έργο των διερμηνέων. γιατί στα Ιταλικά ειδικά πολλές φορές τρώμε τα λόγια μας, είναι δύσκολο για τους διερμηνείς. Τώρα ο Φιλίπ Λαμπέρ έχει το λόγο από τους Πρασίνους. Καλώς ήρθατε στο Κοινοβούλιο. Στην Ιταλία, ε, η Ιταλία δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζεται καλά από το διεθνή τύπο, αλλά σκεφτόμαστε τη χώρα σας. Όταν σκεφτόμαστε τη χώρα σας έχουμε θετικές εικόνες στο μυαλό. Στην Ιταλία οι πολίτες ε, μαζικά εκφράστηκαν υπέρ του να μείνει η ίδρυυση δημόσια υπηρεσία. Στην Ιταλία εκφράστηκαν μαζικά υπέρ της ε, κατάργησης της πυρηνική ενέργεια. Στην Ιταλία δημιουργήθηκε το κίνημα για το slow food, που είναι αντίδοτο στην ταχυφαγία που καταστρέφει, τα στομάχια μα και τι κοινωνίε μα. Και στην Ιταλία, χάρη στον ιστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργήθηκαν 3, εκατομμύρια πράσινων θέσεων εργασία. Όμω η κυβέρνησή σα, κύριε Κόντε, κάνει διαφορετικά πράγματα. Και μα θυμίζει τι χειρότερε στιγμέ που γνώρισε η πυρό μα ορισμένε φορέ. Όταν ο Υπουργό των Εσωτερικών που μοιάζει να είναι ο πραγματικός, ε, το πραγματικό αφεντικό λέει ότι το όνειρό του είναι να απελαθούν οι Ρώμα από τη χώρα σα. Αυτοί που ζουν εκεί. Και επίση η χώρα σα ε, θίγεται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή και μπορεί να αντιμετωπίσει και ύφεση. Και όπω ε, δείξατε και στην ομιλία σας, αποφεύγετε την ευκαιρία να κάνετε την οικολογική μετάβαση, την κινητήρια δύναμη τη οικονομία σα και την κινητήρια δύναμη τη Ευρώπη. Θα μπορούσατε να επιλέξετε να ακούσετε τη, αυτούς που κρούν το κόσμο του κινδύνου, όπως είναι η κυρία Μουρώνη, ή τους δημάρχους που είναι κατά των, κερδοσκοπιών, το... όπως η Ματήλτε Κάζα. Αλλά επειδή θέλετε να υπάρχει μια ξέφρενη ανάπτυξη, ξεκινάτε φαρανονικά και ανόητα προγράμματα, όπως το τούνελ της ε, κοιλάδας του Χιούζ ή της, ε, του περαιτέρου τσιμεντόματος της χώρας από τις της Ευρώπης αντιμετωπίζεται επίση μια δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση. Και εάν βεβαίω φέρουν και οι προκάτοχοί σα ένα μεγάλο ποσοστό τη ευθύνη, κανεί δεν μπορεί να αρνηθεί το ότι η Ιταλία εφήγει από τι πολιτικέ λιτότητε που υπάρχουν μετά τη συνθήκη του Μαστρίχτ. Αλλά αντί να επιδιώξετε να δημιουργήσετε συμμαχίε για να μεταρρυθμίσετε την Ευρωζώνη, του ώστε το κοινό μα νόμισμα να ωφελεί όλα τα κράτη-μέλη, η κυβέρνησή σα τι επιλέγει, αντιπαράθεση ε, δραματοποιεί την κατάσταση, αλλά αυτό δεν οδηγεί σε τίποτα καλό και αυξάνει του κινδύνου. Επίση η χώρα σα είναι στην πρώτη γραμμή τη αντιμετώπιση του ασύλου και τη μετανάστευση. Θα μπορούσατε για την αξιοπρέπεια και την αποφασιστικότητα του Πιέρ του Μπάρτολο να είναι παράδειγμα. Είναι ο γιατρό στην Λαπεντούζα ή του Ντομένικο Λουγκάνο που είναι ο δήμαρχος του Ριάτσε. Θα μπορούσατε να εμπνευστείτε από αυτούς. Αλλά αντί γι' αυτό η του ντομενικο λουγκανο που ειναι ο Δήμαρχο του ριατσε θα μπορουσατε να εμπνευστειτε απο αυτού αλλα αντι γι αυτο η κυβερνηση σα θεωρεί ότι φταίνε οι μετανάστε ε, για όλα τα δεινά τη Ιταλία και κλείνει την πόρτα στα καράβια που σώζουν την τιμή τη Ευρώπη ε, σώζοντα πρόσφυγε. Θα μπορούσατε να δράξετε το απλωμένο χέρι του Κοινοβουλίου που με πολύ ευρία πλειοψηφία ενέχνε την εγκατάλειψη των κανόνων του Δουβλίνου υπέρ τη Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη που και εσεί και η κυβέρνησή σα ε, απαιτείτε. Διότι η μεταρρύθμιση που ενέχνε το Κοινοβουλίο μα ανταποκρίνεται ακριβώ στι απαιτήσει τη κυβέρνησή σα. Αλλά και εδώ το Τσίνκο Εστέλε αντιπαρατέθηκε εδώ κατά την ψηφοφορία. Ενώ η Λέγκα κρύφτηκε πίσω από την αποχή. Αντί γι' αυτό η κυβέρνησή σα προσπαθεί, αντί γι' αυτό, προτιμά αντί γι' αυτό, να συμμαχίσει με αυτού που είναι υπέρ του φρουρίου Ευρώπη, ενώ εγκαταλείπουν την Ευρώπη στην τύχη τη. Και ναι, μεν, ε, το μεταναστευτικό είναι βέβαια θέμα για την Ιταλία. Είναι θέμα για την Ιταλία. Αλλά Υπάρχουν δύο εκατομμύρια νέοι Ιταλοί, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεταναστεύσει ελεύθερα ή υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα του τα τελευταία 15 χρόνια. Πιστεύετε πραγματικά ότι οι αντιφαντικέ και συγκεκριμένε πολιτικέ τη κυβέρνηση θα τους ε, παρακινήσουν να επανέλθουν ή θα σταματήσουν την περαιτέρω διαρροή. Θεωρούμε ότι αν η Ιταλία γίνει κινητήρια δύναμη μιας ε, μετάβασης δημοκρατικής, ε, πράσινης και αλληλέγγυες θα δώσετε ένα μέλλον στη χώρα σας που είναι ανάλογο τη ιστορία τη ανάλογο τη θέση που έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά μας θα είμαστε εκείνοι που θα κινητοποιηθούμε γύρω από αυτές τις προτεραιότητε, κάνοντας έκκληση ε, ε επίγουσες για την Ιταλία. Ευχαριστώ πολύ. Για την Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας το λόγο έχει κυρία Ατζέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε Κατάρινεν, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι η 17η συζήτηση που κάνουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Υπάρχει κίνδυνος να, ενώ όσο συζητούμε για το μέλλον της Ευρώπης, να μην έχει παρόν η Ευρώπη. Εμείς συνεχίζουμε να θεωρούμε την Ευρώπη που ιδρύσαμε ως το σπίτι μας, αλλά η Ένωση χρειάζεται μια βαθιά μεταρρύθμιση γιατί οικοδομήθηκε από την στέγη ξεχνώντας τα θεμέλια. Εμείς θέλουμε να δώσουμε στο σπίτι αυτό στέρεα και διαρκή και δυνατά θεμέλια. Θέλουμε μια Ευρώπη πιο δίκαιοι, πιο σωστοί, πιο κοντά στους πολίτες, χωρίς να υπάρχουν ε, χώρες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Θέλουμε να κερδίσει η πραγματική οικονομία την πρώτη θέση σε σχέση με τη χρηματοοικονομική προσέγγιση. Θέλουμε επενδύσεις, ε, ανάπτυξη, όχι λιτότητα. Θέλουμε μια Ευρώπη που να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και να μην υποκύπτει στις μεγάλες δυνάμεις όπως η Ρωσία, η Κίνα και η ΕΠΑ. Θέλουμε μια ένωση όχι με όνομα αλλά στην πράξη. Και σας ρωτώ, αυτό σημαίνει να είμαστε υπέρ κατά της Ευρώπης. Πολλοί κοιτούν την ε, Ευρώπη, δεν ε, ε, βλέπουν το, την καμπούρα στην πράξη των άλλων, αλλά δεν βλέπουν τη δική τους. Πρώτα χτυπάνε την Ευρώπη και μετά αναγνωρίζουν ότι έκαναν μεγάλο, την Ελλάδα και μετά αναγνωρίζουν ότι έκαναν ένα μεγάλο λάθος. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να σημαίνει να αφήνουμε μια χώρα μόνο να διαχειρίζεται τη μετανάστευση. Το να είσαι ευρωπαϊστή σημαίνει να, δημι... να μετατρέψει φορολογικό παράδοσο... παράδεισο τη χώρα σου. Σημαίνει να αντιμετωπίζουμε σαν ε, πολεμική πράξη την εισαγωγή στην Ιταλία του, ε, ε, του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που αφορά όλη την Ευρώπη. Αυτοί είναι ψεύδο Ευρωπαίοι που έφτιαξαν μια Ευρώπη όχι των πολιτών αλλά των τραπεζών, της γραφειοκρατίας και της λιτότητας μακριά από τους πολίτες. Μπορούμε να αλλάξουμε και πρέπει να μιμηθούμε την Ιταλία που αλλάζει αυτή τη στιγμή. Σε 7 μήνες καταργήσαμε τις ισόβιες προσόδους των ε, παλιών, βουλευτών, κόψαμε τις χρυσές συντάξεις, μειώσαμε τη φορολογία για τις μικρές επιχειρήσεις, ξεκινήσαμε να πληρώνουμε 30 δισεκατομμύρια χρέη των, του δημοσίου στους επιχειρηματίες. Σήμερα στην Ιταλία υπάρχει ε, ε, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Διαλύσαμε τη μεταρρύθμιση των συντάξεων που μας είχε επιβάλει η Ευρώπη για να έχουμε ε, σωστά νούμερα. Κύριε Κατάιν, εγώ είμαι από την Ούμπρια. Μιλήστε για την Όρτσια. Στην Όρτσια το μόνο που χρησιμοποιούνταν είναι να παίρνουν τα χρήματα των επενδύσεων για να τα μοιράζονται μεταξύ τους. Αυτό υποστήριξαμε στους πολίτες και αυτό κάναμε. Εμείς αυτό που λέμε το κάνουμε. Η πρόσφατη έκθεση για το 2019 για την Ιταλία που δημοσίευσε το Εουρίστες, γνωστό ίδρυμα, υπογραμμίζει την αύξηση της εμπιστοσύνης των Ιταλών προς την κυβέρνηση. 15 με 20 ε, ποσοστιαίες ονάδες πιο πάνω. Είμαστε μια κυβέρνηση αλλαγής, ακούμε τους πολίτες και τους παρέχουμε μια νέα ελπίδα για το μέλλον. Γι' αυτό μας κατηγορούν για λαϊκιστές. Κύριε Πρωθυπουργέ, όπως θυμήσατε, αν αυτό σημαίνει να ακούμε τους, ε, να, αυτό σημαίνει να ακούμε τον κόσμο, ναι, είμαστε λαϊκιστές. Δυστυχώς, πολύ συχνά σε αυτό το κτίριο, κτισμένοι στα, κλεισμένοι στα κλουβιά μας, ξεχνάμε να ακούμε τον, τους πολίτες. Ξεκινώντας από την κατάργηση της διπλής έδρας του Κοινοβουλίου, η δομή του, του χώρου στον οποίο είμαστε τώρα, που ερχόμαστε τέσσερις ε, μέρες το μήνα και κοστίζει 200 εκατομμύρια. Εμείς είμαστε φίλοι των Γάλλων και δεν επιτρέπω σε οποιονδήποτε να μας δίνει μαθήματα για, την, για υποστήριξη σε ε, μπαχαλάκιδες. Εμείς δεν δεχόμαστε ότι μπορεί αυτό να θεωρείται αρνητικό. Εμείς δεν λέμε όχι στη δημοκρατία επειδή λέμε όχι στις δύο έδρες. Δεν, δεν σημαίνει όχι στη δημοκρατία γιατί είμαστε κατά ε, των δαπανών που κάνει το Κοινοβούλιο. Θέλουμε να μειωθούν οι τεράστιοι μισθοί των επιτρόπων που είναι πραγματικά κόλαφος για τους πολίτες. Για τις προνομιακές ε, συντάξεις των Ευρωβουλευτών έχουμε ήδη υποβάλει μια πρωτοβουλία. Κύριε Ταγιάννη, υποστηρίξτε την πρότασή μας. Όλα αυτά δεν έγιναν μέχρι τώρα, θα τα κάνουμε εμείς, όμως χάρη στην ψήφο των πολιτών στις επόμενες ευρωεκλογέ και με την συνεργασία των άλλων δυνάμεων της αλλαγής. Έχουμε βάλει στην, ε, στο τιμόνι της Ιταλίας μια πολύ καλή ομάδα τιμονιέριδων. Αυτό θα κάνουμε και στην Ευρώπη σε λίγο καιρό αλλάζουμε την Ιταλία, θα αλλάξουμε την Ευρώπη. Λοιπόν, προς γενική σας πληροφόρηση, θα ήθελα να σας πω ότι η επιλογή της έδρας δεν είναι αρμοδιότητας αυτού του σώματος ή των κρατών μελών που προσυπέγραψαν μια συνθήκη. Λοιπόν, κυρία Ατζέα, θα ήθελα να σας πω ότι εγώ δεν δέχτηκα τις 500.000 που μου προτάθηκαν στα πλαίσια της συνταξιοδότησης και δίνω αυτά τα χρήματα σε μία ομάδα αποτοξίνωσης ναρκωμανών. Η κυρία Πιτζότο, σήμερα κύριε Κόντε μας μιλάτε για την πρώτη πραγματική κυβέρνηση αλλαγών της Ευρώπης που με υπερηφάνεια μιλά για την εθνική μας κυριαρχία. Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Έχουμε ε, το θάρρος να πούμε όχι στις Βρυξέλλες και στα προστάγματα του Βερολίνου. Δεν είμαστε υπέρ του μικρού Ναπολέοντα Μακρόν. Μια κυβέρνηση που υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Ιταλών. Αυτούς τους μήνες η κυβέρνηση Λέγκα Πέντε Αστεριών έδειξε ότι η αλλαγή είναι δυνατή. Ο Ματέο ε, ο Ματέο Σαλβίνη μπόρεσε να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση και αντιμετωπίζουμε και την παράνομη μετανάστευση με την λεγόμενη κότα τσέντο προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε σωστά το συνταξιοδατικό. Πολλά έχουν γίνει κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Να αυτονομηθεί το Βένετο, η Λομβαρδία, η Εμίλια Ρωμάνια, να γίνει μία μεγάλη φορολογική αναθεώρηση, να περικοπούν οι φόροι. Ο Μαδούρο είναι ένας μεγάλος δικτάτορας και είμαστε υπέρ με το λαό της Βενεζουέλας, Βενεζουέλας που θέλει την ελευθερία. Εμείς ήδη εργαζόμαστε, γιατί μετά την Ιταλία θέλουμε να αλλάξουμε από την κορυφή προς τα κάτω ολόκληρη την Ευρώπη και θα το κάνουμε με τη συνένεση του Ιταλικού λαού στις ευρωεκλογές. Η Λέγκα του Σαλβίνη θα γίνει το πρώτο κόμμα της Ιταλίας και το πρώτο κόμμα ολόκληρης της Ευρώπης. Ε, δεν θα είμαστε σκλάβοι των τραπεζών και των πολιεθνικών, των spread και της λιτότητας. Τέλος στην Ευρώπη του Γιούνκερ, της Μέρκελ και του Μακρόν που θέλουν να ταπεινώνουν τους λαούς και το λαό της Ιταλίας. Στην Ιταλία το λόγο έχουν οι Ιταλοί πολίτες, όχι η Μέρκελ ή ο Μακρόν. Μετά τις ευρωεκλογές θα έχουμε την δύναμη να δημιουργήσουμε μια νέα Ευρώπη, την Ευρώπη των λαών της ελευθερίας, της υπεράσπισης των συνόρων, του Made in Italy, της ε, αναχέτησης των μεταναστών στα σύνορά μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, νομίζουμε ότι η κυβέρνησή μας θα διαρκέσει για πολύ, θα είναι για πολύ στην εξουσία, γιατί έχουμε μία αποστολή να υπερασπιστούμε τη γη μας από τους γραφειοκράτες των Βρυξελών και να υπερασπιστούμε την εθνική κυριαρχία. Μπράβο σας κύριε Πρωθυπουργέ. Γουλφ από τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε Πρωθυπουργέ Κόντε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ σήμερα. Κύριε Πρωθυπουργέ της Ιταλίας, η αποφασιστικότητα της κυβέρνησής σας να αντισταθεί στη, στα, στην προνομιακή πρόσβαση στην εξουσία της Μέρκελ και του Μακρόν και να αντισταθεί στις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελίτ που είναι εδώ παρούσες και προτείνουν ότι η κυβέρνησή σας είναι ρατσιστική, φασιστική και ότι είναι ανδρίκελα του Πούτιν και ότι είναι αντιφεμινιστική και αντιευρωπαϊκή. Σας χειροκροτώ για την δράση σας. Εσείς εμπνέετε τους δημοκράτες παντού στην Ήπειρο και στον κόσμο. Η κυβέρνησή σας έχει καταδείξει ότι η Ευρώπη δεν είναι αυτός ο θεσμός που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι είναι ένας, ε, μία ήπειρος αρχαίων λαών, αρχαίων εθνών. Αρχαίων λαών, αλλά με σύγχρονες μεθόδους. Ορισμένες φορές φοράνε κίτρινα γυλαίκα. Ορισμένες φορές ψηφίζουν Brexit. Ορισμένες, όπως οι συνάδελφοί σας από τα πέντε αστέρια, χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα και τα κάνουν πολιτική εξουσία για τους ε, απλούς ανθρώπους. Είναι σύγχρονες οι μέθοδοι για αρχαίες φωνές, αλλά οι φωνές αυτές πρέπει να εισακουστούν. Η συζήτηση σήμερα αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς και η κυβέρνησή σας και οι συναδελφοί σας είστε το μέλλον της Ευρώπης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στον Πρωθυπουργό της Ιταλικής Δημοκρατίας για να απαντήσει στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Μετά έχουμε το Catch the Eye. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα θέματα που θίξατε είναι πολυπίκυλα κινούμαστε από θέματα ευρωπαϊκού αποτυπώματος σε θέματα που αφορούν την εθνική μας πολιτική, την πολιτική της Ιταλικής Δημοκρατίας. Θα αρχίσω από ένα θέμα που θίξατε, θα ομαδοποιήσω στις απαντήσεις μου και θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα θέμα που απασχόλησε σχεδόν όλους, ε, την μετανάστευση. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Θα ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω ότι αυτό που έκανε η κυβέρνησή μου συγκεκριμένα ήταν να δει την πραγματικότητα κατάματα. Ο καθένας μπορεί να αντλήσει τα συμπεράσματά του, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα γεγονότα καθεαυτά. Από την πρώτη στιγμή αυτής της ε, πολιορκίας γνωρίζουμε βέβαια ότι η μετανάστευση οδηγεί σε διχογνωμίες και τη στιγμή που είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες ελιμενισμούς δεν είχαμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές γιατί λόγω της γεωγραφικής μας ε, θέσης, μερικοί το ξεχνάτε, αλλά είμαστε στην καρδιά της Μεσογείου και από την ε, κεντρική Αφρική έχουμε άπειρες ροές. Γνωρίζοντας το τι συνέβη και γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτή μία αλόγιστη υποδοχή, γιατί διαφορετικά θα μπορούσε να υπάρχει και ένταξη. Δεν γίνεται ένταξη έτσι. Ένας συνάδελφός μου, ένας πρωθυπουργός ευρωπαϊκής χώρας, είχε αντιμετωπίσει την μετανάστευση από απόσταση. Μετά μου είπε Τζουζέπε, κατανοώ ότι έχετε ένα μεγάλο πρόβλημα όταν έβλεπα στους δρόμους ε, δεκάδες δεκάδες μετανάστες. Πώς το αντιμετωπίσαμε με μία διαρθρωμένη απάντηση. Καταλάβαμε ότι πρόκειται για μία κατεπίγουσα κατάσταση που δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε εύκολα. Ορίσαμε λοιπόν 10 στόχους σε σχέση με την πολιτική, ε, με τις χώρες διαμετακόμισης, από που αρχίζει αυτή η πορεία των μεταναστών, οι χώρες ε, διαμετακόμισης και εδώ μιλώ και για παράκτιες ε, χώρες. Μιλήσαμε λοιπόν για κατανομή αντιμετώπιση και επαναπατρισμούς. Κατά το πρώτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη Ιουνίου, όπου συμμετείχα, μιλήσαμε για αυτά τα συμπεράσματα, φτάσαμε σε αυτά τα συμπεράσματα και μιλήσαμε για κοινέ στοχοθετήσεις και όποιος στην στην ουσία φτάνει στην Ιταλία, φτάνει στην Ευρώπη. Είναι ένα θέμα το οποίο δεχτήκαμε. Έμπρακτα όμως, ακόμα και σήμερα, δεν έχουν βρεθεί λύσεις. Είχαμε πολλά ευρωπαϊκά συμβούλια έκτοτε, αλλά καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια να θέσουμε σε εφαρμογή αυτές τις αρχές. Και δεν φταίει η Ιταλία γι' αυτό. Δεν φταίει η Ιταλία.